η περίοδος συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει διακοπεί και σας εύχομαι σε όλους καλή και ασφαλή επιστροφή και ωραίο Σαββατοκύριακο.